Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ο Μάρκ Ρόζερσον. Η εκλογική εκστρατεία έχει λήξει. Έχουν ψηφίσει οι πολίτες. Η δημοκρατική διαδικασία έλαβε χώρα. Πάνω από 150 κανάλια στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένα μαζί μας για να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα. Θα σα δώσουμε τα στοιχεία τη προσέλευση σε όλη την Ευρώπη, τα πρώτα στοιχεία για τα αποτελέσματα και μια εικόνα για την πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου. Και θα ακούσουμε και τι απόψει των πολιτικών ηγετών τη Ευρώπη. Στο Βερολίνο, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans-Gerd Pöttering. Στι Βρυξέλλε, μαζί μα ο Ζωζεφ Ντόλ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Στο Βερολίνο επίση ο Μάρτιν Σούλτ, ο πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πράσινους, ο συμπρόεδρος τους, ο Ντανιέλ Κομπεντίτ, θα είναι στο στούντιό μας στο Παρίσι και ήδη στο Παρίσι είναι ο Φρανσίς Βίρτς, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστερά. Σε λίγα λεφτά οι δημοσιογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στους πολιτικούς. Αλλά ας ξεκινήσουμε με μερικά στοιχεία για το θέμα της προσέλευσης και τη συμμετοχή των πολιτών, ο Ζαμιντού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας παρουσιάσει. Ο Ζαμιντούτς, σε ευχαριστώ. Θα σας δώσω κάποιες εκτιμήσεις που περάσουμε στα αποτελέσματα, τις ε, εκτιμήσεις για τη συμμετοχή των πολιτών. Και για τη συμμετοχή και για τα αποτελέσματα βασιζόμαστε σε εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων TNS χρησιμοποιώντας πραγματικά αποτελέσματα αλλά και εν μέρη ε, με τα exit polls. Τώρα θα ήθελα να παρουσιάσετε το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό για την Ευρώπη στα 27 κράτη-μέλη. Euh, λοιπόν, 43,39% η συνολική συμμετοχή των πολιτών στις εκλογέ. 1% λιγότερο από ότι το ποσοστό του 2004 και του 2007. Και τώρα οι προβλέψεις για τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς δεν είναι οριστικά αποτελέσματα. Υπάρχουν ψαλίδες που δείχνουν το προβλεπόμενο αριθμό εδρών και σιγά σιγά θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. Η τελευταία λοιπόν πρόβλεψη είναι ως εξή για τα κόμματα σε σχέση με την ε, προβλεπόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 263 με 273 έδρες. Σοσιαλιστική ομάδα 155 με 165 έδρες. Οι φιλελεύθεροι και δημοκράτες 78 με 84 έδρες. Η πράσινη και ελεύθερη συμμαχία 52 με 56 έδρες. Η Γκουε 33 με 37 έδρες, ενωτική αριστερά δηλαδή, η Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών 33 με 37 έδρες, η Ανεξαρτησία Δημοκρατία 15 με 19 έδρες και 83 με 89 έδρες ακόμα οι οποίες κατανέμονται στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ενδεχομένω θα δημιουργηθούν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα λοιπόν όπως τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Γυρίζω το λόγο στον ε, και πρέπει να σας πω ότι είναι παρόν μαζί μας ο Γκραμ Γότσον από τον ε, Συνεσπισμό Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Πάμε όμως τώρα στο Βερολίνο όπου είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Hans Gert Böttering. Πώς βλέπετε τα αποτελέσματα κυρία Böttering και ιδίω το μελλοντικό σχήμα, η μελλοντική σύνθεση του Κοινοβουλίου. Ποια θα είναι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συμμετέσχαν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι αυτό το ποσοστό συμμετοχής θα μπορούσε να ήταν υψηλότερο και θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο τα επερχόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των <clears throat> βουλευτών από τα κόμματα και των μέσων ενημέρωσης. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με μεγάλη φροντίδα θα πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι στο μέλλον. Με μεγάλη χαρά καταγράφω το γεγονός ότι τα ευρωπαϊστικά κόμματα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι έχουν πράγματι αποκομίσει μια μεγάλη ευρωπαϊστική πλειοψηφία και γι' αυτό θέλω να κάνω και μια έκκληση να βασιστούμε σε μια κοινή δράση των ευρωεπαριστικών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε την οικοδόμηση της Ευρώπης και περιμένω από τα κόμματα τα οποία δεν έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ένα δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω και να συγχαρώ όλους αυτούς οι οποίοι εξελέγησαν στο νέο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Πέτριν. Στις Βρυξέλλες έχουμε τον Ζωζεφ Τόλ, ο είναι ο πρόεδρος του ΕΛΚ και έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε τη δική σας άποψη. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκλογείς, τους ψηφοφόρους που ακολούθησαν το μήνυμά μας, τις γυναίκες, τους άντρες, το ΕΛΚ που δούλεψαν πολύ επί τόπου πάνω στα διάφορα θέματα που προωθούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ψηφοφόρους μας και πράγματι όταν βλέπει κανείς τα νούμερα για το ΕΛΚ Βέβαια και είμαι ικανοποιημένο. Βλέπω ότι με διαφορά κερδίσαμε και ότι οι σοσιαλιστές κάπως έχασαν σήμερα το βράδυ. Um, ναι, Βερολίνο τώρα. Για να απαντήσει στο σχόλιο του Ζώσεφ Ντόλ. Ο Μάρτιν Σούλτ, λοιπόν, πρόεδρος των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mr. can you hear me? Μ' ακούτε, κύριε Σούλτς, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ωραία. Μήπω θέλετε να σχολιάσετε τα αποτελέσματα και τις προβλέψει που έχουμε ως στιγμής. Ναι, σίγουρα είναι πολύ λυπηρή η βραδιά αυτή για τι ισοδημοκρατίε στην Ευρώπη. Απογοητευθήκαμε πάρα πολύ. Ελπίζαμε σε καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ορισμένα κρατημένα λυπήκαν τα πράγματα για μας πολύ καλά, στα περισσότερα όμως πολύ άσχημα. Και υποφέραμε το γεγονό ότι ε, είχαμε σημαντικότητα σε είτε σε ορισμένε χώρε λόγω της εσωτερικής πολιτικής των κρατών αυτών. Γενικά είναι πικρή η απόψινή βραδιά για μας. θα προτιμούσα να σχολιάσω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά στη δημοκρατία πρέπει κανένας να αποδεχθεί αυτό που του προσφέρουν οι ψηφοφόροι. Τα θέματα μας ξεκολουθούν να παραμένουν επίκαιρα. Η κοινωνική Ευρώπη είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη σήμερα, ακόμα περισσότερο απαραίτητε είναι οι σε χρηματοπιστωτικές αγορές, περισσότερο επίση η προστασία του κλίματος, η ε, παρεμπόδιση του αν, της ανεξάρτητης εξέλιξης ε, του καπιταλισμού θα προσπαθήσουμε πάση θητεία να επιβάλλουμε την κοινωνική μας ε, ατζέντα. Θα έχουμε τελικά 180 περίπου έδρες, ίσως και κάτι παραπάνω και με αυτά επίσης μπορεί κανένας να εργαστεί πολύ καλά. Ευχαριστώ. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να παραδώ τον Γκρέμ Βότσον. Τι έχετε να πείτε μέχρι απόψε. Δεν έχουμε ακόμα όλα τα αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ότι η φιλελεύθερη ομάδα θα επανέλθει στο νέο κοινοβούλιο με την ίδια ισχύ όπως το προηγούμενο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να ε, μπορούμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ της εράς και της δεξιάς. Θα είμαστε ισχύς που θα συμβάλλει στο αποτέλεσμα των περισσότερων ε, ψηφοφοριών και θα εξακολουθούμε να είμαστε μια υπερευρωπαϊκή δύναμη στο κέντρο του σώματος. Τα αποτελέσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά χαίρομαι που μπορέσαμε να προχωρήσουμε ως φιλελευθέροι στην Ευρώπη. Γενικά η συμμετοχή είναι χαμηλή. Καμία από τις ομάδες δεν φαίνεται ότι ενθουσίασαν τους ε, ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, είμαστε κάπως προσεκτικοί στη χώρα μου ε, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ υψηλή όταν οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι. Είναι δικαίωμα των πολιτών η ψήφος. Μπορούν να αποφασίσουν θα ξέρουν. Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω. Θα ήθελα να φροντίσουμε όλοι οι ε, επίτροποι να ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, να έχουμε ένα ποσοστό των ε, ευρωβουλευτών σε κοινά ευρωπαϊκά ε, ψηφοδέλτια και επίσης οι δημοσιογράφοι να παρουσιάσουν τα θέματα κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ο Ντάνιελ Κόνμπεν δεν έχει φτάσει ακόμα στο Παρίσι. Θα περάσουμε λοιπόν στον Φράνσις Βίρτς που είναι στο στούδιο. Τι έχετε να μας πείτε για τις εξελίξεις μέχρι στιγμής. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι το ποσοστό αποχής που αυξήθηκε πρέπει όλους να μας κινητοποιήσει, να μας κάνει να ανησυχήσουμε, γιατί δείχνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης από πάρα πολλούς πολίτες απέναντι στην Ευρώπη έτσι όπως αυτή οικοδομείται σήμερα. Έπειτα, από αυτούς που πήγαν στις κάλπες και ψήφισαν, το βάρος της δεξιάς είναι και το βάρος των ξενοφοβιστικών δυνάμεων, των λακιστικών δυνάμεων, γιατί προς το παρόν εμείς οι δυνάμεις της αριστεράς και άλλοι δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του κόσμου. Όσον αφορά τη δικιά μου πολιτική οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, αν λάβουμε υπόψη μας το ότι ο αριθμός των εδρών έτσι κι αλλιώς μειώνεται, από 49 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σχετικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς παραμένει λίγο πολύ σταθερό σε διάφορες χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και άλλες. Προδεύουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά την Ιταλία. Δεν ξέρω. Γενικά πάντως πιστεύω ότι κρατάμε το σχετικό μας βάρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να δουλέψουμε όχι τόσο βάσει του πνεύματος στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέτερινγκ, τον οποίο εκτιμάω ιδιαίτερα και σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του εδώ. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης και είμαι ιδιαίτερα επικριτικός στους σημερινούς προσανατολισμούς της Ευρώπης. Με γνωρίζει ο κύριος Πέτριν καλά και καταλαβαίνει πολύ καλά και το ξέρει ότι μπορεί κανείς να είναι υπέρ της Ευρώπης αλλά να κατακρίνει τους σημερινούς προσανατολισμούς της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι σήμερα η Ευρώπη δεν βαδίζει καλά. Ευχαριστούμε, Φρανσίς Βούρτς. Ο Ντάνιελ Πετίτ σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας. Οπότε, η προεκλογική αυτή εκστρατεία είναι μια εκστρατεία που έχουν παρακολουθήσει χιλιάδε δημοσιογράφοι μέσα στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτού βρίσκονται εδώ στο ημικύκλιο αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τι ερωτήσει του προ του πολιτικού ηγέτε. Ο Τζαουμέ Ντού έχει το λόγο, εκπρόσωπο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Μάρκ. Λοιπόν, όποιο θέλει το λόγο να σηκώνει το χέρι του και όταν του δίνουμε το λόγο να ρωτάτε στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα γερμανικά τι ερωτήσει σα να πείτε και ποιοι είσαστε και σε ποιον πρόεδρο ομάδος ή στον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται την ερώτησή σας. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Με την πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Σηκωθείτε για να σας βλέπουμε καλύτερα. Ποιος θα ξεκινήσει? Λυπάμαι, αλλά δεν βλέπουμε κανέναν. Α, εδώ έχουμε μία ερώτηση. Παρακαλώ. Γαλλικά, αγγλικά ή γερμανικά την ερώτησή σας, παρακαλώ. Στην Ιταλία ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι ο ορισμός του επόμενου Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας Ιταλός, ο Μάριο Μάουρο, και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Όσον αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 Ιουλίου θα τον ψηφίσουμε. Σήμερα είμαστε εδώ με δύο υποψήφιους από πλευράς του ΕΛΚΑ, ο Μάριο Μάουρο και ο κύριος Μπούσεκ από την Πολωνία και μαζί έχουμε συζητήσει τη συζήτηση αυτή για τον πρόεδρο να την κάνουμε μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Από αύριο δηλαδή. Θα δούμε αν υπάρχει λύση. Αν δεν υπάρχει, η δημοκρατία θα αποφασίσει. Ξέρετε ότι όταν ήμουν εγώ υποψήφιος είχαμε τέσσερις υποψηφίους. Ε, η δημοκρατία κατέληξε, έβγαλε το αποτέλεσμα. Η συζήτηση πάντως θα ξεκινήσει από αύριο για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ο Σάιμον. Να πάει το μικρόφωνο μια στιγμή. Σάιμον Τέιλερ από την European Voice. Μια ερώτηση προς τον κύριο Σούλς παρακαλώ. Γιατί πιστεύετε ότι η σοσιαλιστική ομάδα τα πήγε τόσο άσχημα. Περιμένατε 200 έδρες, οπότε φαντάζομαι και τότε λέγατε ότι θα, θα ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα τώρα. Ε, τι έχετε να πείτε, φταίει οικονομική κρίση. Äh, Είδαμε ότι σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποτελέσματα ήταν πολύ διαφορετικά. Πάλι ορισμένα από εξελίξεις της εσωτερικής πολιτικής και σκέψεις για την εσωτερική πολιτική των ψηφοφόρων. Η σοσιαλιστική ομάδα είχε γι' αυτό ένα κακό αποτέλεσμα γιατί διάφορα από τα κόμματα μας τα ε, διάφορα κράτη-μέλη είχαν κακό αποτέλεσμα και στη δία μου τη χώρα. Θα ήταν καλό λοιπόν τις επόμενες μέρες να εξετάσουμε σε κάθε χώρα γιατί υπήρξε το αποτέλεσμα που υπήρχε. Θα πρέπει να εξετάσουμε το αποτέλεσμα στη Μεγάλη Βρετανία πολύ προσεκτικά, στη Γερμανία προσεκτικά, το ίδιο για τη Γαλλία και για κάθε χώρα θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ ειδικοί λόγοι στην εκάστοτε χώρα που δεν είχαν καμία σχέση παραπάνω περιπτωριακά με την εργασία της ε, κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Αυτή είναι η εξήγηση που έχω να σα δώσω. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Udo van Kampen, Από το ZF Udo van Kampen, μια ερώτηση προς τον κύριο Watson. Εάν οι φιλελεύθεροι μαζί με τους σοσιαλιστές προσπαθήσετε να αποτρέψετε μια επανεκλογή του κυρίου Περόζο. Με συγχωρείτε, σας βλέπω. Ωραία. Θα πρέπει καταρχήν να οργανώσουμε την ομάδα μας και μετά να αποφασίσουμε. Εμείς προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ομάδα για τη δυνατότητα μιας ιδεολογικής, δηλαδή πολιτικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Είμαστε κατά μιας νέας ε, τεχνικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων πολιτικών ομάδων. Η Ευρώπη οι, συμπολίτε οι συμπολίτες μας αποφασίσανε στις κάλπες για κάποιο συγκεκριμένο κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίσουμε το αποτέλεσμα αυτό και να δημιουργήσουμε μια ιδεολογική ένωση, έναν ιδεολογικό συνασπισμό εδώ στο σώμα. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου συμφωνεί μαζί μου για το θέμα αυτό. Ε, το επόμενο ερώτημα. Σηκωθείτε παρακαλώ για να σας δω. Από την Σουηδική τηλεόραση προς όλους τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων πόσο χαμηλή μπορεί να φτάσει να είναι η συμμετοχή των εκλογέων ώστε να σας κάνει να θέλετε τα εθνικά κοινοβούλια να εκλέγουν τους ευρωβουλευτές πλέον και όχι ο λαός. Ο κύριος ε, Πέτρος στο Βερολίνο. Θέλετε να απαντήσετε. Δεν το άκουσα πολύ καλά από την, ε, από την απόσταση. Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημά σας. Με το μικρόφωνο αυτή τη φορά. Προσπαθήσω να σας το, να το πω στα γερμανικά, από τη σουηδική τηλεόραση. Πόσο χαμηλή πρέπει να είναι η εκλογική συμμετοχή ώστε να είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε στο προηγούμενο σύστημα όπου οι ευρωβουλευτές εκλέγονται από τα εθνικά κοινοβούλια. Μα πρέπει να σας πω, λέει ο πρόεδρος Πέτεριν, ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω το ερώτημα αυτό. Είναι βέβαια σημαντικό να αυξηθεί η εκλογική συμμετοχή των πολιτών. Αλλά το να θέλουμε τα, Ευρω... εθνικά κοινοβούλια να εκλέγουν τους ευρωβουλευτές, αυτό το απορρίπτωσαν σαν θέση. Εγώ είπα προηγουμένως ότι οι βουλευτές, τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης και στα οποία ανήκει και ο ερωτών θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα πρέπει καλύτερα να παρουσιάσουν την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών, αυτό όχι μόνο πριν από τις εκλογές και κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, αλλά σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή τη βελτίωση και θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι έγινε σαφές σε μένα την προηγούμενη εβδομάδα ότι όταν γίνεται η ανανέωση του, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου της ε, Γερουσίας τα τελευταία 35 χρόνια η συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις εκλογές ήταν κάτω από 40%. Δεν το λέω για να το θεωρήσουμε σαν παράδειγμα, απλώς σας το υπενθυμίζω. Ο στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι η πολιτική υπεύθυνη και τα μέσα ενημέρωση τα οποία ανήκετε και εσείς να εξασφαλίσουμε στα επόμενα πέντε χρόνια ότι οι ειδήσει και η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι σωστή και συνεχής γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο και επομένως και οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα για να έχουμε το 2014 καλύτερη εκλογική συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντόλ, θέλετε και εσείς να πείτε κάτι. Όχι. Γιατί θα έλεγα ακριβώ τα ίδια πράγματα που είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι είναι γεγονός ότι πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τα Εθνικά Κοινοβούλια ως ΕΛΚ εδώ και δύο μισή χρόνια έχουμε αποδηθεί σε μια στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και να την κάνουμε στενότερη. Το πρόβλημα όμως το οποίο τίθεται και το είδα στην προεκλογική εκστρατεία είναι ότι οι εθνικοί βουλευτές δεν γνωρίζουν ποια είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αποφασίσουν οι υπουργοί τους στις Βρυξέλλες θα πρέπει να ενημερώνονται και αυτοί για τα θέματα αυτά στις εθνικές ε, επιτροπές των ε, κοινοβουλίων. Αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ο κύριος Σούλτς τώρα από το Βερολίνο. Παρακαλώ. Θέλετε και εσείς να δώσετε την απόψή σας. Τα είπε όλα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, όλα αυτά τα οποία έπρεπε να πει κάποιος και νομίζω δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ένα μικρό σημείο μονάχα λέει ο Γκραχαμ Βότσον. Δεν ξέρω, πρέπει να το μελετήσουμε καλύτερα γιατί δεν κατεβαίνουν στις κάλπες οι πολίτες και δεν ψηφίζουν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουν κάποια σύνδεση μεταξύ της πολιτικής έκφρασής τους στην ψηφοφορία, της ψήφου τους και της μορφής της διακυβέρνησης των θεσμών της Ευρώπης για τις οποίες ψηφίζουν. Νομίζω ότι αν υπήρχε μια φέστερη σύνδεση μεταξύ της ψήφου και του αποτελέσματο με τη μορφή της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ή τη δημιουργία μιας πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψήφισαν περισσότεροι πολίτες. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εκλέγονται ορισμένοι σε πανευρωπαϊκές λίστες για να υπάρχει πραγματικά ευρωπαϊκή συζήτηση και να ζητούμε από το Συμβούλιο να επιλέγει τους υποψηφίους τους από αυτούς που εκλέγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της θέλησης των πολιτών και της εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βίρτς έχει το λόγο. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς τους ευρωβουλευτές έκανε την προεκλογική του εκστρατεία, όπως και εγώ. Συναντηθήκαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας μίλησε κανείς για ποιο τρόπο εκλέγουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι. Αυτό που έρχεται στη συζήτηση είναι η πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικυρώνεται από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε την ιδέα ότι η ελευθέρωση αυτή των ε, κοινοφελών υπηρεσιών, αυτός ο ανταγωνισμός, ο ακραίος, αυτή η ανεργία που μας πλήττει είναι πράγματα τα οποία δεν περνάνε πια. Ο κόσμος όταν δεν βλέπει προοπτική μπροστά του λέει «Ε τότε γιατί να πάω να ψηφίσω αφού τελικά η πολιτική φαίνει ίδια». Πάτε το γαλλικό παράδειγμα. Πριν από τέσσερα χρόνια υπήρξε μια πλειοψηφία κατά της συνταγματικής ε, συνθήκης, όχι γιατί ήταν κατά της Ευρώπης, αλλά ήταν κατά των ε, φιλελεύθερων ιδεών της Ευρώπης αυτής. Ε, και τι έγινε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρήκε τον τρόπο να εγκριθεί τελικά η συνθήκη της Λισαβόνας που ουσιαστικά είναι μια λίγο αλλαγμένη μορφή της δαγματικής συνθήκης αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Οπότε ο κόσμος λέει «Ε τι νόημα έχει να πάω να ψηφίσω, ας κάτσω σπίτι μου καλύτερα». Ε, λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε τελικά τι πολιτική κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για το πώς χειριζόμαστε και πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα. Ευχαριστούμε κύριε Βίρτς. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Ράδιο Πούντο, Ράδιο Ρανέ. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στους άλλους πρόεδρους. Σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, να ο κύριος Βούρτ αναφέρθηκε σε αυτήν. Λοιπόν, τώρα με τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι θα γίνει. Η συνθήκη αυτή θα εγκριθεί και αν δεν εγκριθεί, τι θα γίνει. Τι μέλη γενέστε. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτή και να σας πω ότι είχε συμφωνηθεί ότι θα είχαμε 35 λεπτά για το συζήτηση αυτή. Έχουμε και άλλες υποχρεώσεις και σας παρακαλώ δείξτε ε, κατανόηση ότι θα πρέπει να τηρήσουμε και τις άλλες μας υποχρεώσεις. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Η συνθήκη της Λισαβόνης είναι μία συνθήκη πάνω στην οποία εργαστήκαμε 10 χρόνια μαζί με τη συνταγματική συνθήκη. Από τότε δηλαδή που ενεκρίθη η συνθήκη της Νίκαιας, Δεκέμβριο 2000. Και η συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά πιο ικανή να δρά την Ευρωπαϊκή Ενόμαση, να είναι πιο δημοκρατική και πιο διαφανής και θα εκμεταλλευτώ κάθε δυνατότητα που έχω για να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη αυτή γιατί τη χρειαζόμαστε για να υπάρχει ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Ζητόρ, νομίζω θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσει το λιγότερο δυνατό να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Αφώνας. Θα περιμένουμε βέβαια πρώτα τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας και κάποιες υπογραφές από κάποιες χώρες αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τεθεί σε ισχύ και θα έχει και περισσότερες αρμοδιότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το εξηγήσαμε στη δημοκρατική μας, ε, ε, στην προεκλογική μας εκστρατεία ότι μας ρωτάνε τι κάνουμε, ποιες είναι αρμοδιότητες. Ξέρετε κύριε Βίρτς, συνεργαστήκαμε πολύ καλά, αλλά εάν οι Γάλλοι ήταν πράγματι κατά της Ευρώπης, όπως αφήνεται να ερωθεί και γι' αυτό δεν ψηφίζουν νομίζω τον αντίον θα είχαν πάει να ψηφίσουν για να καταψηφίσουν την Ευρώπη γιατί για πρώτη φορά είχαμε εκείνους που ψήφισαν υπέρ της Ευρώπης γιατί όλη μου η εκστρατεία ήταν ε, βασισμένη στην εργασία που ε, επιτελέσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια που σκοπεύουμε να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια γιατί πραγματικά συνεργαστήκαμε και με τη Γαλλική Προεδρία για τα μεγάλα θέματα. Υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να βρούμε από κοινού από την κρίση αυτή στην Ευρώπη. 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Είναι σημαντικό αυτό. και περιμένουν οι πολίτες συγκεκριμένες λύσεις για να βγούμε από το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι απελπισμένοι, έχετε δίκη. Αλλά τώρα θα προτείνουμε όμω μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία για να βγούμε από την κρίση αυτή. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει. Ευχαριστώ κύριε Ντόλ. Ξέρω ότι ορισμένοι από του προσκεκλημένου μα πρέπει πολύ γρήγορα να φύγουν. Αυτό που θα κάνω θα δώσω τη δυνατότητα και στον κύριο Σούλ, στον κύριο Βότσον και στον κύριο Βέρτς να απαντήσουν και μετά θα κλείσει αυτό το τμήμα της συνέντευξης τύπου. Κύριε Σούλτς, παρακαλώ. Εγώ ελπίζω ότι θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Το έργο που έπρεπε να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ πιο εύκολα βάσει της συνθήκη της παρά βάσει της συνθήκη τη Νικιάς. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή σα σε κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα απόψε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, ένα από τα πιο ισχυρά σώματα του διεθνούς κοινοβουλευτισμού. Αποφασίζουμε για νομούς που ισχύουν για τους πολίτες 27 χώρες μέλη. Όταν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας θα συμπεριληφθούν αλλά οι 80 περίπου τομεί πολιτική όπως παραδείγματος κάνει και η αγροτική πολιτική, μέσα στα πλαίσια των αρθμοδοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό. Εάν όμως από την άλλη μεριά, όσο πάει γίνεται πιο ισχυρό το Κοινοβούλιο και ταυτόχρονα μειώνεται η συμμετοχή στι εκλογές, και οι εκλογές αυτές στα κράτη-μέλη, όπως και σήμερα, δεν, έχει δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική της Ευρώπης. Δεν νομίζω η Μεγάλη Βρετανία ψηφίσει σαν για την ευρωπαϊκή πολιτική, ούτε στην Ουγγαρία, για να δώσουν αυτά τα δύο παραδείγματα. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα έγιναν πολύ περισσότερο από εκείνα που φανταζόμαστε έτσι εκ πρώτης ματιά θα πρέπει να συζητήσουμε, βρισκόμαστε σε μια κρίση νομιμότητας. Η ερώτηση του Σουηδού δημοσιογράφου, στην οποία απάντησε σωστά ο κύριος Πέτερινγκ, δείχνει όμως ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα για την επανεθνικοποίηση της Ευρώπης. Η ερώτηση αυτή έδειξε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το ότι το θέμα της νομιμότητας βάση των εκλογών και της συμμετοχής των εκλογών θα πρέπει να προωθηθεί. Αν δεν το καταφέρουμε θα έχουμε πολύ σκληρούς καιρούς μπροστά μου. Εγώ θα προσπαθήσω με τα, τις λίγες δυνατότητες που έχω ως ε, βουλευτής να συμβάλλω στην επόμενη θητεία για το αυτό. Κύριε Σουότσον. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα αν ίσχυε η συνθήκη της Λισαβόνης. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις συνθήκες. Τους ενδιαφέρει η δουλειά που γίνεται. Ε, θα δουλέψει. Και αν δείτε τι έγινε το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς ε, που πέρασε τον Αύγουστο, κινητοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για να κρατεθούν τα ρωσικά στρατεύματα έξω από την Τυφλίδα. Το ίδιο κινητοποιηθήκαμε και για τις τράπεζές μας. Τον ε, Νοεμβρίο, τον Δεκέμβριο κινητοποιηθήκαμε ώστε να έχουμε καλή πολιτική για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αυτά θέλει να δει ο κόσμος. Και αν τους πείσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει, τότε θα είναι πιο ευτυχής και θα πάνε να υπερψηφίσουν τη συνθήκη της Λισαβόνας που μας δίνει τις εξουσίες που θέλουμε. Παρακαλώ, κύριε Υπάρχει μια παρεξήγηση κάθε φορά που μιλάμε για ευρωπαϊκέ συνθήκε, συμπεριλαμβανομένε και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Για μια μεριά υπάρχει το θεσμικό θέμα, οι εξουσίε και αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν είμαι κατά τη αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι τη συνθήκη τη Λισαβόνα που αυτό δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Είναι το οικονομικό και το κοινωνικό φιλελεύθερο μοντέλο. Τις πρόλες άκουσα ή μάλλον διάβασα δηλώσει του Προέδρου του Eurogroup, του Jean-Claude Juncker, που έλεγε ο ίδιος προσοχή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί πάμε προς μια μεγάλη συζήτηση για το οικονομικό και κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Και η συζήτηση αυτή θα οδηγήσει σε έκρηξη. Ε, περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε απλώς να λέμε «Α, πρέπει να επικυρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η συνθήκη της Λισαβόνας». Πρέπει να ξέρουμε, στη σημερινή συνθήκη, όπως και σε εκείνη της Λισαβόνας, τι δημιουργεί πρόβλημα στους Ευρωπαίους πολίτες και γι' αυτό απομακρύνονται από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο με λυπεί βαθύτατα, γιατί ό,τι και νομίζει ο κύριος Ζωζεφ Ντόλ, εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης. Πρέπει να ανοίξει λοιπόν αυτή η συζήτηση, να γίνει, ορισμένοι τη φοβούνται, αλλά πρέπει να γίνει πιο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο θέλει η πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Και αν πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση, ε, να το κάνουμε, να δεχτούμε αυτή την αλλαγή. Αν θέλουμε και πάλι να βρεθούμε πιο κοντά στους πολίτες οι οποίοι απομακρύνονται από εμά όπως βλέπουμε. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θέλει να παρέμβει για να κλείσουμε αυτήν τη συνέντευξη τύπου. Αλλιώς νομίζω θα δώσουμε τέλος στη συνέντευξη τύπου. Ναι, θα ήθελα μια ακόμα φορά να λάβω το λόγο για να ευχαριστήσω τους πολίτες που έχουν ψηφίσει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ευρία πλειοψηφία υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και ζητώ από τα κόμματα να συνεργαστούν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τον δρόμο για να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο ευρωπαϊκό χώρο για την πολιτική και αυτό είναι θέμα και των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη και των πολιτικών οικογενειών να αναζητήσουν λύσεις μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητώ και από τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν την πρέπουσα θέση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αξίζει μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και τις καλύτερες μου ευχές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Τα σχόλια του Πρόεδρου Πότερινγκ μας έφεραν στο τέλος της ειδική μετάδοσης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προτού κλείσουμε να σας υπενθυμίσω ποια είναι η πιθανότερη μορφή του νέου Κοινοβουλίου. Πρέπει να βάλω και τα γυαλιά μου γιατί είναι σε μια οθόνη που δεν βλέπω πολύ καλά. Η Γκουε Βόρεια Αριστερά 33 με 37, οι Σοσιαλιστές 155 με 165, οι Πράσινοι 52 με 56, ο συνασπισμός φιλελευθέρων και μεταρρυθμιστών 78 με 84, το ΕΛΚ 263 με 273. Α, έχω την εικόνα. Η Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών 33 με 37 έδρες, Ανεξαρτησία Δημοκρατία 15 με 19 και οι υπόλοιπε έδρες είναι 83 και 89. Θα είναι ένα ενδιαφέρον κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολιτικούς ηγέτες εδώ στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στο Παρίσι και ευχαριστούμε την τεχνική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έκανε δυνατή αυτή τη μετάδοση σε όλη την Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόντες εδώ απόψε. Καλό βράδυ.